Καλό απόγευμα σε όλους και όλες. Θα αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Το πρώτο σημείο της ημερησίας διατάξεως είναι η έγκριση της ημερησίας διάταξης. Θα ήθελα να σας προτείνω δύο αλλαγές. Η πρώτη σχετίζεται με την έκθεση κυρίας Νέντελ Σέβα το σημείο 13 δηλαδή, ζήτησε να ε, ψηφιστεί αύριο η έκθεσή της γιατί πρέπει να συμμετάσχει σε μια άλλη συνεδρίαση. Δεύτερη αλλαγή σε σχέση με την έκθεση της κυρίας Βένσον δεν μπορεί να παραστεί στη συνεδρίαση αυτή τη βδομάδα και ζητάει να γίνει ψηφοφορία για την έκθεσή της, να αναβληθεί μάλλον η συζήτηση για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, να αφαιρεθεί δηλαδή από το σχέδιο μερίσιας διάταξης ε, της σημερινής συνεδρίασης και να αναβληθεί η συζήτηση για την επόμενη συνεδρίαση. Αυτό είναι το σημείο 15. Αν ε, δεν υπάρχουν ενστάσεις, εγκρίνουμε το σχέδιο μερίσιας διάταξης ούτως τροποποιημένο. Σημείο 2. Ανακοινώσεις ε, της Προέδρου. Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση υπό αυτό το σημείο. Περνούμε στο σημείο 3 έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων των 8 ε, Νοεμβρίου και 29 έως 30 Νοεμβρίου 2010. Έχουμε μοιράσει ήδη τα πρακτικά. Αν μέχρι το πέρας της τωρινής συνεδρίασης δεν προκύψει κάποια ένσταση, θα θεωρήσω ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο 4, το πλέον σημαντικό σημείο της σημερινής μας συνεδρίασης. Πρόκειται για την παρουσίαση του προγράμματος της Ουγγρικής Προεδρίας για τον δικό μας ε, τομέα, δηλαδή ισότητα των φίλων και δικαιώματα των γυναικών. Ο Υπουργό Εθνικών Πόρων της Ουγγαρίας, ο κύριος Μικλός Ρέτελη, είναι μαζί μας. Τον καλωσορίζω και θα του δώσουμε απευθείας το λόγο για να ακούσουμε την παρουσίαση του προγράμματος της Ουγγρικής Προεδρίας για το τρέχον εξάμεινο ως προς τα θέματα που μας αφορούν, δηλαδή την ισότητα των δύο φίλων και τα δικαιώματα των γυναικών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κυρία Ρέτελη. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι βουλευτές, με μεγάλη μου χαρά έρχομαι στη σημερινή σας συνεδρίαση για να παρουσιάσω το πρόγραμμα της Προεδρίας μας ε, και να εκθέσω τις προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας για το τρέχον εξάμεινο. Θα σας εξηγήσω ακριβώς πώς θα προωθήσουμε τα θέματα, ε, της πρωτοβουλίες ε, που άπτονται της ισότητας των δύο φύλων. Υπάρχουν ε, σχετικά χαμηλές προσδοκίες, διότι προσχώρησε η χώρα μας ε, πριν από έξι χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα περασμένα έξι χρόνια η Ουγγαρία αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση βίωσαν σημαντικότατες αλλαγές. Η συνθήκη της ε, Λισαβόνας προσέδωσε στο Κοινοβούλιο επιπρόσθετες αρμοδιότητες και συνιστά ένα νέο έρισμα για τις σχέσεις ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Είμαι πεπισμένος ότι θα έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου και ευελπιστώ ότι θα κατορθώσουμε να βρούμε απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα ε, που για τα οποία μάλλον θα πρέπει να ληφθούν κοινέ αποφάσεις. Για τις ε, γυναίκες ε, έχουν σημειωθεί πολύ σημαντικέ αλλαγέ τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μια, ας αρχίσουμε μια θετική αλλαγή. Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών αυξήθηκε σημαντικά. Μέσα σε μία δεκαετία, από το 1998 μέχρι το 2008, σημειώθηκε αύξηση άνω του 7%. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ε, στοιχείο που οφείλουμε να λάβουμε υπόψη εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικότερε διαφορές στα ποσοστά ανασχόληση αντρών και γυναικών αντίστοιχα. Το 2008 η διαφορά, η ποσοστιαία διαφορά ανερχόταν σε σχεδόν 14%. τι ούτω τρόπος οι μισθολογικές διαφορές ανάμεσα στους ε, άντρες και στις γυναίκες ε, μειώθηκαν. Το ίδιο ισχύει για το κίνδυνο ε, φτώχειας και για τη θέση των γυναικών και αντρών στην κοινωνία. Βεβαίως δεν ήταν τόσο σημαντικές οι αλλαγές που σημειώθηκαν όσο είχαμε υπολογίσει αρχικά και ε, επιπροσθέτως ε, στις επιμέρους περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ισχύουν τα ίδια δεδομένα. Τώρα με την χρηματοοικονομική κρίση είδαμε ε, σημαντικές επιπτώσεις οι οποίες όμως διαφέρουν ε, ανάλογα με το αν εξετάζουμε την κατάσταση των αντρών ή των γυναικών. Δηλαδή, ε, γυναίκες που έχασαν τη θέση αποσχόλησης του δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας και μετά από μία μακρά περίοδο ανεργίας αναγκάστηκαν να ε, δεχτούν θέσεις ε, που δεν είναι καλά αμοιβόμενε και χαρακτηρίζονται από κακές συνθήκες εργασίας. Τώρα, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουμε να ρίξουμε τα θεμέλια της μελλοντική οικονομικής ανάπτυξης. Και η ισότητα των φύλων είναι εκ των όνου κάνευ προϋπόθεση για την αύξηση της απασχόλησης και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε πως είναι προφανές ότι δεν ε, ωφελεί να συζητούμε την ε, στρατηγική Ευρώπη 2020 δίχως να ε, προσδίδουμε την δέουσα έμφαση στη διάσταση της ισότητας των δύο φύλων. Ο ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι η ευφυής βιώσιμη και αλληλέγγυα ανάπτυξη. Ε, δεν δυνάμεθα να επιτύχουμε κανέναν από τους στόχους της στρατηγικής αυτής χωρίς να προσφέρουμε τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες, είτε είναι γυναίκες είτε είναι άντρες, τη δυνατότητα να μετάσχουν σε όλες τις διαδικασίες στα κοινά και να έχουν τα ίδια ωφέλη από την ανάπτυξη. Ω προ την ισότητα των δύο φύλων τώρα, αυτό το θέμα είναι πολυδιάστατο. Έχουμε τι εμβληματικέ πρωτοβουλίε πρωτοβουλίες, υπονομαζόμενες flagship initiatives και εκεί πρέπει να σωματώσουμε και τι δύο διαστάσει τη ισότητας των δύο φύλων. Γιατί πράγμα σα μιλώ για τη συμφιλίωση καταρχά ανάμεσα στην ιδιωτική ε, και την επαγγελματική ζωή, την αναβάθμιση των συνθήκων εργασία ε, των γυναικών και την ενίσχυση του ρόλου του στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Γιατί αναφέρομαι πρώτα απ' όλα στην στρατηγική Ευρώπη 2020, διότι η εφαρμογή της αρχίζει ε, κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Προφανώς όλες οι σχετικές πρωτοβουλίες υπάγονται στις αρμοδιότητές μας. Στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ θέλουμε να ασχοληθούμε όλος ιδιαίτερως με την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την πρόθεση της ένταξης των Ρωμά. Εάν υπάρχει ε, πολιτική βούληση εκ μέρους όλων και αν υπάρχει συνοχή στο έργο μας, τότε η δημιουργία θέσεων απασχόλησης θα μπορούσε να μας βοηθήσει να μειώσουμε τις ανισότητες των δύο στην αγορά εργασίας Αντίστοιχα, μιλώντας τώρα για την ένταξη των Ρωμά, οι δράσεις μας θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ε, διαβίωση και την οικονομική κατάσταση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων καθώς και να προωθήσει να ενισχύσει το ρόλο των γυναικών Ρωμά στην κοινωνία. Υφίστανται και άλλες δύο βασικές προκλήσεις, η δημογραφικές τάσεις ε, στην Ευρώπη και ε, προφανώς το φαινόμενο της γύρανσης ε, του πληθυσμού συνεπάγεται μεγάλες προκλήσεις. Για να αντεπεξέλθουμε σε αυτές τις προκλήσεις, οφείλουμε να επιτύχουμε μια ισορροπία. Γιατί συμφιλίωση, όπως έλεγα, της ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, πρώτα απ' όλα θεωρούμε ότι είναι εφικτό να συμφιλειωθεί η προσωπική και η επαγγελματική ζωή και αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για το θέμα της ισότητας των δύο φύλων. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η φροντίδα μιας οικογένειας ε, ταυτόχρονα με την εργασία αφορά πολύ περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άντρες. Στην πράξη αυτό σημαίνει διπλό φόρτο εργασίας ε, για τις γυναίκες για αυτούς τους λόγους ε, υφίστανται διακριτική μεταχείριση πολύ περισσότερες γυναίκες από ότι άντρες ε, στην αγορά εργασίας. Και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να επιληφθεί του ζητήματος ε, η Ουγγρική Προεδρία και θα ρίξουμε νέο φως σε αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζοντας τις δημογραφικές προκλήσεις στην Ευρώπη. Η στρατηγική Ευρώπη 2020 έχει θέσει ε, ε, λίγα φιλόδοξους ε, στόχους, οι οποίοι όμως δεν θα επιτευχθούν εάν δεν καταφέρουμε να ανταποκριθούμε με ορθό τρόπο σε αυτές τις νέες προκλήσεις του δυναμικού της αγοράς εργασίας, εάν δεν καταφέρουμε να αντεπεξέλθουμε στις δημογραφικές προκλήσεις. Για να αποφύγουμε η αδίποτε παρανόηση, θα ήθελα να τονίσω και κάτι άλλο. Η Ουγγρική Προεδρία πιστεύει ότι πέρα από την στρατηγική Ευρώπη 2020, πιστεύει λοιπόν ότι όλε οι διαστάσει του ζητήματο τη ισότητα των δύο φύλων είναι εξίσου σημαντικέ και θα πρέπει να μα απασχολούν ε, με πάγιο τρόπο. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να μην χειριζόμαστε αυτά τα ζητήματα και ταυτόχρονα να ισχυριζόμαστε ότι προαγάγουμε την ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι κατά τη διάρκεια ενό εξαμήνου είναι ανέφικτο να καλύψουμε όλα τα ζητήματα και όλες τις ε, εκφάνσεις, όλες τις ε, ε, διαστάσεις ενός ζητήματος. Και δεν θα πρέπει λοιπόν να πέσουμε στην παγίδα του να έχουμε υπερβολικά φιλόδοξους στόχους και τελικά να έχουμε μηδαμινά αποτελέσματα. Επιλέξαμε λοιπόν τρεις προτεραιότητες που σχετίζονται με τα δικαιώματα των γυναικών και το θέμα της ισότητας των δύο φύλων. Υπάρχουν χιλιάδες ζητήματα συναφή, αλλά εμείς επιλέξαμε τρεις προτεραιότητες. Είναι οι εξής. Πρώτον, θέλουμε να αναθεωρήσουμε το θέμα της ισότητας των δύο φύλων υπό το φως της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Δεύτερον, θέλουμε να τονίσουμε την επιτακτική ανάγκη της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών και τρίτον θα θέλαμε να προωθήσουμε εν γέννη την ισότητα των δύο φύλων, διατομεακά δηλαδή. Ε, προφανώς ε, δεν είναι ιεραρχημένες αυτές οι προτεραιότητες ως προς τη σημασία τους, ε, τις ε, ανέφερα μόνο επιγραμματικά είναι όλες εξίσου σημαντικές και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ε, λεπτά ε, ακαθόδη ζητήματα ε, που σχετίζονται με συγκεκριμένους τομείς, αλλά δεν τα έχουμε συμπεριλάβει στο πρόγραμμά μας. Επίσης θέλουμε να προωθήσουμε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την ε, Ισότητα των Δύο Φύλων που εγκρίθηκε το 2006 και να ε, βασιστούμε ε, σε αυτό για τις εργασίες μας. Γιατί χρειάζεται λοιπόν να προωθήσουμε αυτό το σύμφωνο. Για μια σειρά λόγων και πάλι εδώ επιγραμματικά, επιγραμματικά θα παριθμίσω τους λόγους. Πρώτον, χρειαζόμαστε, χρειάζεται αναθεώρηση αυτού του συμφώνου διότι από την έγκρισή του και μετά έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές ε, στις ε, οικονομίες και στις κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και με κάποιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και να προσαρμοστούμε στις αλλαγές. Δεύτερον, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να λάβουμε δεόντως υπόψη τα απ τα αποτελέσματα με την εφαρμογή αυτού του συμφώνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το θέμα της ισότητας των δύο φύλων και τρίτων. Η Στρατηγική Ευρώπη 2020 έχει δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο συγγνώμη, για την οικονομική ανάπτυξη, ένα οριζόντιο πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να γίνει σεβαστό και τέλος εξίσου σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη στρατηγική της για τα δύο φύλλα για την περίοδο από το 2010 έως το 2015. Το Συμβούλιο Ε, μέσα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ καλωσόρισε το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε αυτά τα συμπεράσματα αναφέρεται ε, συγκεκριμένα η αναθεώρηση του Συμφώνου ισότητας των Δύο Φύλων. Τι εισηγείται λοιπόν η Ουγγρική Προεδρία για την μεταξέλιξη, αν θέλετε, αυτού του Συμφώνου. Θα θέλαμε να προσδιορίσουμε πρώτα απ' όλα ένα χρονοδιάγραμμα για να διευκολύνουμε έτσι και την παρακολούθηση της εφαρμογής του Συμφώνου. Πιστεύουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε με πλέον αποτελεσματικό τρόπο να συμβάλλουμε στην εφαρμογή της ε, Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Του τέστη θα θέλαμε να ορίσουμε τις προτεραιότητες και τις πολιτικές μας ε, δεσμεύσεις ε, για την ίδια αυτή περίοδο ως προς το θέμα της ισότητας των δύο φύλων. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι ε, θα έχουμε προτεραιότητες και δράσεις για την εφαρμογή των οποίων χρειάζεται περίοδος μακρύτερη της ε, δεκαετίας. Ε, παρόλα αυτά ε, θα ήταν χρήσιμο για όλους πιστεύουμε να χρησιμοποιούνται οι ίδιες βασικές αρχές, το ίδιο χρονοδιάγραμμα και η ίδια ιεράρχηση προτεραιοτήτων όταν εφαρμόζουμε το σύμφωνο. Παρά την έγκρισή του το 2006 παραμένει επίκαιρο το σύμφωνο από πολλές πλευρές διότι όπως σας εξήγησα ήδη παρά τις προσπάθειες που έγιναν εξακολουθεί να υπάρχει ένα χάσμα ε, ανάμεσα, ε, μια ε, πολύ σοβαρή μισθολογική διαφορά ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες, σοβαρή διακριτική μεταχείριση στην αγορά εργασίας. Δεν έχουμε επιτύχει δηλαδή τους στόχους μας και αναφέρομαι μόνο σε κάποιους επιμέρους στόχους του συμφώνου. Ε, υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα στοιχεία του τωρινού συμφώνου που θα θέλαμε να παραμείνουν μετά την αναθεώρηση, Θα οποία όμως δεν θα αναφερθώ τώρα. Ταυτόχρονα Είναι σημαντικό να αναφερθούμε στην επιτακτική ανάγκη καταπολέμησης της βίας που υφίστανται οι γυναίκες. Αυτό έλειπε από το σύμφωνο του 2006. Ε, παρά το φαινόμενα που παρατηρούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι προηγούμενε προεδρίε ε, ήδη επέστησαν την προσοχή όλων στην έλλειψη αυτή του συμφώνου. Και συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια. Πρόκειται για, μια, για, για τη σοβαρότερη παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών. Αν δείτε τα αριθμητικά στοιχεία, σίγουρα θα θελήσετε να αναλάβετε δράση. Τουλάχιστον δύο στις δέκα γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πέσει θύμα ε, βίας ε, και κυρίως σεξουαλικής βίας, ασέλγειας, κακοποίηση. Ε, δεν θα μπορέσουμε βέβαια να χειριστούμε όλες τις ε, λεπτομέρειες ε, του προβλήματος, αλλά προφανώς μπορούμε να προσδιορίσουμε γενικούς στρατηγικούς στόχους. Γι' αυτό το λόγο θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη που θα εκπονήσουν τις στρατηγικές τους, να εισηγηθούν ένα πλαίσιο για την έγκριση δράσεων και πολιτικών αποφάσεων κατά όλων των μορφών βίας που υφίστανται οι γυναίκες. Ταυτόχρονα θέλουμε να τονίσουμε τον σημαντικότατο ρόλο που διαδραματίζουν οι άντρες ε, στην καταπολέμηση της ε, βίας ε, κατά των γυναικών. Χαίρομαι όλους ιδιαίτερος διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πάγιο τρόπο πραγματεύεται αυτό το θέμα στις διάφορες επιτροπές και το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει, επεξεργάζεται μια άλλη συμφωνία που θα αποτελέσει επίσης ε, σημαντικό βήμα προόδου. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια ανταλλαγή εμπειριών, να συλλέξουμε όλες ε, τις εμπειρίες ε, των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, διότι μέσω της συλλογής των εμπειριών θα εμπνευστούμε για το μελλοντικό μας έργο. Βέβαια, όλες αυτές ε, οι προθέσεις ε, πρέπει να μεταφραστούν σε δράσεις, σε ενέργειες και χρειαζόμαστε και περισσότερη παρακολούθηση των ε, δράσεων. Γι' αυτό θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην υλοποίηση και στην παρακολούθηση, εποπτεία. Ελπίζουμε ότι έτσι κάθε κράτος μέλος θα τονίσει περισσότερο αυτά τα θέματα της ε, διάστασης του φύλου και της ισότητας μεταξύ των ε, φύλων όπως είναι στην Ατζέντα 2020 και στα εθνικά προγράμματα. Τώρα, ας συνεχίσω με δύο πολύ ευαίσθητους νομοθετικούς φακέλους οι οποίοι είναι το οι εξής. Είναι σημαντικοί φάκελοι. Πρώτον, η οριζόντια ε, οδηγία κατά των διακρίσεων και δεύτερον, η οδηγία για την ε, ε, άδεια λοχίας. Άδεια, μητρό, άδεια γονική, άδεια τοκετού. Λοχίας μάλλον. Ε, θα πρέπει λοιπόν να βρεθούμε σε, σε μια δύσκολη κατάσταση όταν θα προσπαθήσουμε να υιοθετήσουμε και να, να εγκρίνουμε τις λεπτομέρειες των δύο αυτών οδηγιών. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις στα κράτη-μέλη όσον αφορά την υλοποίηση, την εφαρμογή των διατάξεων. Και αυτό γιατί συμβαίνει, διότι διαφέρει η πρακτική εφαρμογή των δύο αυτών τομέων στα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να ε, προσπαθήσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Άλλωστε μας ε, χαρακτηρίζει το γεγονός ότι είμαστε ενωμένοι μέσα σε πολλές διαφορετικότητες. Τώρα βέβαια δεν χρειάζεται να τονίσω πόσο σημαντική είναι η οδηγία κατά των διακρίσεων. Η υιοθέτηση μιας τέτοιας οδηγίας θα συμπληρώσει ε, τα κενά ε, του νομοθετικού πλαισίου που υπάρχουν σήμερα, τα κενά της ελλείψης. Διότι όσον αφορά την αποφυγή των διακρίσεων, οι διάφορες ενέργειες που γίνονται σήμερα είναι διαφορετικές και βασίζονται ε, στο, στα αίτια της, ε, των διακρίσεων. Για, ποιο λόγο δηλαδή γίνονται αυτές οι διακρίσεις. Δεν θα πρέπει λοιπόν να διαφοροποιήσουμε στην εφαρμογή ανάλογα με τα αιτία, ανάλογα με την πηγή και για ποιο λόγο γίνονται οι διακρίσεις. Θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον εξασφαλίσει ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας κατά των διακρίσεων. Ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμείς έχουμε συμφωνήσει να προωθήσουμε κοινά ε, κοινού στόχους και κοινέ αξίες και να συντονίσουμε τις ενέργειές μας, τις δράσεις μας σε ορισμένους τομείς. Όσον αφορά το, αυτή την οδηγία λοιπόν κατά των διακρίσεων, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ε, με μία οριζόντια οδηγία η οποία δεν ε, κινείται μέσα στα πλαίσια της αγοράς, των αγορών μάλλον. Δεν μπορούμε να σας δώσουμε καμία υπόσχεση για το πότε θα ολοκληρωθεί αυτός ο φάκελος. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία σε αυτό το θέμα με το σημερινό οικονομικό δυσμενές κλίμα. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι θα χειριστούμε με πνεύμα ισότητας, με μια ίση προσέγγιση όλες τις οδηγίες οι οποίες περιλαμβάνουν το στοιχείο της, των διακρίσεων. Η Ουγγρική Προεδρία έχει στα χέρια της λίγα, αλλά θέλουμε να καταφέρουμε πολλά. Θέλουμε να Εστιάσουμε επίσης την προσοχή μας στην προστασία των ατόπων με ειδικέ ανάγκες. Αυτό το θέμα είναι μια συνέχεια της Βελγικής Προεδρίας, αλλά δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο ε, διαλέξαμε ε, την εστίασή μας σε αυτό το θέμα είναι μία προτεραιότητα στο πλαίσιο της διάστασης των φύλων για την ε, Ουγγρική Προεδρία και έχει άμεση σχέση με τις διαβουλεύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ατόμων με ειδικέ Ανάγκες, το European Disability Strategy. Θέλουμε λοιπόν να επιτύχουμε συνέργεια και γι' αυτό αποφασίσαμε να προτείνουμε μέτρα τα οποία θα εγγυώνται προστασία ε, σε άτομα τα οποία έχουν ειδικέ ανάγκες. Είναι σαφώς θέμα και αυτό ε, διακρίσεων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό θα οργανώσουμε ε, μια διάσκεψη ψηλού επίπεδου και το αντικείμενο θα είναι η εδραίωση ενός νομοθετικού πλαισίου ε, ευρωπαϊκά και διεθνώς. Πιστεύουμε ότι η συναφής ε, σύμβαση του, των, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πρέπει να επικυρωθεί το συντομότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήμασταν ευτυχής να δεχθούμε και μέλη της Επιτροπής σας ε, ε, ως συμμετέχοντες δηλαδή σε αυτό το συνέδριο. Πολλές φορές έχουμε μιλήσει υπέρ της τήρησης ορισμένων αρχών, όμως πολλές φορές πραγματικότητα είναι διαφορετική, είναι σκληρή. Το γεγονός είναι ότι έχουμε έναν κατάλογο προτεραιοτήτων, όμως λόγω των μεγάλων διαφορών που υπάρχουν πρέπει να βρούμε ένα συμβιβασμό. Πρέπει να βοηθήσουμε να προστατεύσουμε τις έγκυες γυναίκες, πρέπει να προστατεύσουμε το ε, έμβριο, πρέπει να προστατεύσουμε ε, τη διαδικασία του τοκετού, πρέπει να προστατεύσουμε την κοίηση, τον τοκετό και τη λοχεία όλες τις φάσεις. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα συμφέροντα ε, των ε, εργοδοτών και τις ανάγκες της αγοράς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αγνοήσουμε ε, τους ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν μια οικογένεια. Επίσης πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις δημογραφικές τάσεις. Η Ουγγρική Προεδρία δεν έχει καμία, κανέναν ενδιασμό να ασχοληθεί με αυτά τα καυτά θέματα. Χρειαζόμαστε, όπως σας είπα, ελάχιστα, ελάχιστες απαιτήσει, ελάχιστα standards σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διαφορές των κρατών μελών για να καταλήξουμε σε ελάχιστα standards. Τώρα, όσον αφορά την άδεια τοκετού και λοχείας, εδώ το θέμα είναι πολύ περίπλοκο. Το ξέρουμε αυτό. Η πιο σημαντική διαφορά μεταξύ των κρατών μελών είναι η διάρκεια. Η διάρκεια και η αποζημίωση που λαμβάνει, η χρηματική τυχόν αποζημίωση που λαμβάνει η Λεχόνα. Θα θέλαμε λοιπόν να απαντήσουμε στις προτάσεις σας και η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου θα τις μελετήσει προσεκτικά. Ε, ακόμα και τις προτάσεις δικές σας που ε, είναι πέραν των προτάσεων της Κομισιόν, ξεπερνούν τις προτάσεις της Κομισιόν. Θα θέλαμε να ξεκινήσει μία επεγγελματική συζήτηση μεταξύ ημών και της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για να μπορέσουμε να δούμε ποιο είναι το περιθώριο λιγμών για να βρούμε ένα συμβιβασμό. Επίσης θα θέλαμε να αναθεωρήσουμε την αρχική πρόταση της Κομισιόν προς το Συμβούλιο. Την αρχική πρόταση. Υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη στο Συμβούλιο που μας έχουν πει ότι θα μπορούσαν ως σημείο κίνησης να λάβουν το, την πρώτη πρόταση της Κομισιόν προς το Συμβούλιο η Ουγγρική Προεδρία είναι φιλόδοξη. Όμως δεν θέλουμε να θέσουμε στόχους που δεν είναι ρεαλιστικοί. Γι' αυτό όσον αφορά την άδεια τοκετού και ελοχία. πιστεύουμε ότι σε δύο μήνες υπό την Προεδρία μας θα μπορέσουμε να επιτύχουμε συμφωνία μέσα στο πλαίσιο της συναπόφασης. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται, έχει ανάγκη αυτής της οδηγίας. Ε, πρέπει να συμφωνήσουμε στο τέλος της ημέρας. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Πιστεύουμε, η Ουγγρική Προεδρία πιστεύει ότι η συζήτηση στο Συμβούλιο θα είναι επικοδομητική, ανοιχτή και διαφανής και τέλος θα ήθελα να σας πω πόσο Είμαι ευτυχής να σας φιλοξενήσω, να σας υποδεχτώ στις 16 Μαρτίου στη Βουδαπέστη. Ευχαριστώ πολύ και είμαι πρόθυμη στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε ε, κύριε Υπουργέ. Ρετέλη. Ήταν διεξοδική η παρουσίασή σας σχολιάσατε μεταξύ άλλων κάποια χάσματα, κάποια κενά που υπήρχαν σε σχέση με το πρόγραμμα της Ουγγρικής Προεδρίας, δηλαδή αναφερθήκατε σημαντικά συγκεκριμένα στην καταπολέμηση της ε, βίας κατά των γυναικών, αναφερθήκατε στην άδεια μητρότητας και στην αύξηση της απασχολησιμότητας ε, των γυναικών. Δηλαδή είναι θέματα που δεν προκύπτουν από το έγγραφο του προγράμματος της Ουγγρικής Προεδρίας. Τώρα βέβαια μας τα εκθέσατε με σαφήνεια. Ε, έχουμε πολλούς βουλευτές στον κατάλογο μιλήτων. Αν συμφωνείτε, θα ήθελα να κάνουμε ένα πρώτο γύρο, να ακούσουμε τους εκπροσώπους όλων των πολιτικών ομάδων, κατόπιν να ακούσουμε τις απαντήσεις του Υπουργού και κατόπιν να ε, προβούμε σε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Αν συμφωνείτε με την προτινόμενη μεθοδολογία θα την ακολουθήσουμε και θα ακούσουμε την κυρία Μπάουερ ε, εξ του ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Υπουργέ, για την ε, παρουσίαση. Καλωσορίζουμε το πρόγραμμα ε, της Προεδρίας σας. Θα ήθελα να θέσω ε, κάποιες ερωτήσεις που σχετίζονται με το πρόγραμμά σας. Η πρώτη σχετίζεται με τη Στρατηγική Ευρώπη 2020. Ε, θεωρούμε ότι υπάρχουν διάφορες αντιφάσεις στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής. Ε, θέλουμε να αυξήσουμε την γεννητικότητα και την απασχολησιμότητα ταυτόχρονα. Και γι' αυτό κρίνω ότι είναι ε, ορθέ οι προτεραιότητε τη Ουγγρική Προεδρία, γιατί ρίχνεται το βάρο στη συμφιλίωση τη προσωπική και επαγγελματική ζωή και υπάρχει ένα νέο στοιχείο που μας εκθέσατε, δηλαδή η αναθεώρηση του Συμφώνου του 2006 για την ισότητα των δύο φύλων. Πρώτη ερώτηση. Έχετε κάποιες συγκεκριμένες ιδέες, προτάσεις για την συμφιλίωση της ε, ιδιωτικής και επαγγελματικής ε, ζωής ε, χωρίς να πληγούν άλλα επιμέρους στοιχεία στρατηγικής και δεύτερον για το σύμφωνο του 2006 αν θυμάμαι καλά, ε, ε, ε, ήταν το πόρισμα ενός τριμερούς διαλόγου που συμμετείχαν και οι κοινωνικοί εταίροι. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Προτίθεστε να ξεκινήσετε νέα διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, ούτω ώστε να καταλήξετε σε ένα αναθεωρημένο κείμενο. Είναι πάρα πολύ καλό που συνδέεται το σύμφωνο με την ε, στρατηγική 2020, διότι για να είμαι ειλικρινής, όπως γνωρίζετε και γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, αυτή λοιπόν η στρατηγική δεν εμπεριέχει καμία αναφορά για πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη ε, η ισότητα των δύο φύλων. Παρότι παρότι από πλευρά ε, της απασχόλησης ή της δημογραφικής πρόκλησης ε, ε, είναι ένα κέριο ζήτημα που οφείλουμε να πραγματευτούμε. Καλωσορίζω λοιπόν την νέα προσέγγιση της Ουγγρικής Προεδρίας, το ότι θέλετε να σχετίσετε το σύμφωνο με τη στρατηγική 2020, να συσχετίσετε το σύμφωνο με τη στρατηγική 2020. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο θα το πετύχετε αυτό. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Η κυρία Τόμψεν τώρα από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την ε, ουσιαστική σας παρέμβαση, εισήγηση. Αναφερθήκατε πολύ συχνά σε θέματα τα οποία υπερβαίνουν το πρόγραμμά σας και που αφορούν την ισότητα των φύλων. Σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε για τη βία κατά των γυναικών, γιατί εγώ πιστεύω ότι η πρωτοβουλία που ελήφθη υπό την Ισπανική και μετά τη Βελγική Προεδρία θα συνεχιστεί υπό την Ουγγρική Προεδρία βία κατά των γυναικών. Είναι ένα τεράστιο και πολύ σοβαρό θέμα στην Ευρώπη. Γιατί βεβαίως άπτεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα να ξέρω εάν έχετε την πρόθεση να υποστηρίξετε την εργασία που κάνουμε τώρα στο Κοινοβούλιο για μία οδηγία πλαίσιο ε, κατά της ε, βίας, ε, για τη βία κατά των γυναικών αν θα υποστηρίξετε αυτή την εργασία. Είπατε επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε τις γυναίκες μέσα στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων. Η λήψη των αποφάσεων περιλαμβάνεται ως στοιχείο στο πρόγραμμα της Κομισιόν 2010-2015 και πολλές κυβερνήσεις επίσης έχουν ασπαστεί αυτό το στόχο η Ισπανική κυβέρνηση ε, ε, έχει, η Ισπανική κυβέρνηση έχει ένα υψηλό ποσοστό γυναικών ε, στην κυβέρνηση επίσης στη Γαλλία η, η κυβέρνηση του πρόεδρου Σαρκοζή στη δικιά μου χώρα ε, όμως εσείς στην Ουγγαρία έχετε μια κυβέρνηση η οποία είναι μόνο άνδρες. μόνο οι άντρε εκπροσωπούνται, το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο, διότι δεν συμφωνεί με αυτά που είπατε. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω εάν η πρόθεση της Προεδρίας είναι να αναλάβει μια πρωτοβουλία που να βοηθήσει και ενισχύσει τις γυναίκες για τη λήψη αποφάσεων. Σας Η κυρία τώρα Σας ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε και για όσα μας εξηγήσατε. Να σας πω κάτι, ότι τουλάχιστον στην πτυχή τη θεωρητική που αναπτύξατε εδώ, όλοι στην Επιτροπή συμφωνούμε. Νομίζω. Αλλά ίσως είμαστε κάπως κουρασμένοι και κουρασμένες να ακούμε συνέχεια θεωρητικά πράγματα. Τι γίνεται, αυτό που μας λείπει είναι κάτι το πιο συγκεκριμένο. Εδώ από όσα άκουσα θέλω περισσότερο, κάτι περισσότερο συγκεκριμένο για συγκεκριμένα στοιχεία ε, πάνω στα οποία θα εργαστεί η Ουγγρική Προεδρία. Και δύο θέματα σημαντικά σχετικά με την ε, μητρική αυτή φροντίδα, όπως είπαμε, τη φύλαξη και μας είπατε ότι όλα αυτά έχουν, ε, είναι γεμάτα προβλήματα. Θα πρέπει να έχουμε κάτι το συγκεκριμένο. Τι θα γίνει, τι θα κάνει η Ουγγρική Προεδρία, γιατί τον αναλύει κανείς να παροτρύνει, να δει και πάλι, να ξαναναλύει όλα αυτά. Είναι πολύ καλό, αλλά χρειάζεται κάτι το συγκεκριμένο. Ποιες δραστηριότητες, ποιες πρωτοβουλίες θα αναλυφθούν και τι θα μπορεί να γίνει ακριβώς κατά τη διάρκεια αυτής της Προεδρίας. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω επίσης και για την ειλικρίνειά σας. Είπατε ότι δεν θα υποσχεθείτε περισσότερα, ξέρετε τις δυνατότητες που υπάρχουν, ξέρετε ποιες δυσκολίες έχουν αυτές οι πρωτοβουλίες και ότι είναι σύντομο το εξάμεινο και σχετικά με τα άτομα με προβλήματα. Εντάξει, ε, τα υποστηρίζω πλήρω γιατί οι γυναίκε με παρόμοια προβλήματα υπόκεινται σε διπλή διάκριση. Αυτοί να αντιμετωπίζουν και σχετικά ακόμα με τις άδειε μητρότητα ή πατρότητα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Μπορείτε να μας πείτε όλα αυτά ε, και τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη ποια είναι και μήπως πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε μια συμφωνία πάνω και με την σύμφωνη άποψη του Κοινοβουλίου. Είπατε ότι αυτές οι διαφορές σχετικά ε, με αυτές τις μητρότητες, μητρότητα μητρότητας και των δύο, τι γίνεται ότι θα πρέπει να τα ε, σεβαστούμε και να έχουμε και μια σφαιρική γενική Ευρώπη σεβόμενη και τις διαφορές. Εδώ παντού βλέπουμε ότι χρειάζεται να σεβαστούμε την ισότητα των δύο φύλων, τη μη διάκριση. Εδώ όμω θα πρέπει να είμαστε πιο οξείς και αυστηροί μπορούμε να πούμε και αυτό θα ήθελα να ζητήσω γιατί από τη στιγμή που λέμε όλοι ότι ναι είναι βασικό θεμελιώδης δικαίωμα χρειάζεται να δώσουμε τη μάχη μας κατά της διάκριση και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές οι πτυχές θα πρέπει να λάβουν συγκεκριμένο χαρακτήρα και ακριβώς εκεί θα πρέπει από τη στιγμή που μιλάμε για παρόμοια δικαιώματα πρέπει να τα φροντίσουμε κιόλας και χρειάζεται να ενσωματωθούν ακόμα στις πρωτοβουλίες αυτές και άνδρες και να μπορέσουμε να χτίσουμε μια πραγματική ισότητα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Τώρα από τους Πρασίνους η κυρία Κορνέλησεν παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σχολιάσω κι εγώ αυτές τις δύο οδηγίες που αναφέρατε. Είπατε κάποια ανησυχητικά πράγματα, κάτε με. Η οδηγία περί άδειας μητρότητας. Ε, εγώ στην πρώτη συζήτηση που έγινε στο Συμβούλιο απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Κάποια κράτη-μέλη συγκεκριμένα είπαν ότι η πρόταση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν μια καλύτερη βάση διαπραγμάτευση. Ειλικρινά εγώ το θεωρώ αυτό προσβλητικό ε, ενώπιον του Κοινοβουλίου. Ε, δεν αναγνωρίζουν ποια είναι η διαδικασία θέσπισης νέων νομοθετημάτων ε, ουσιαστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει την πρωτοβουλία υποβολής ε, του σχεδίου Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς οι αιρετοί, ε, αν θέλετε, τοποθετούμαστε και μεταφέρουμε την άποψη του λαού για αυτή την πρόταση. Και αυτή είναι η βάση μετά για να εγκριθεί το νομοθέτημα και όχι η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με όλο το σεβασμό που τρέφω για σας, πιστεύω ότι θα ε, είναι πάρα πολύ δύσκολε οι διαπραγματεύσεις διαβούλευση στο Συμβούλιο, διότι υπάρχει σοβαρή διάσταση απόψεων ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Πάντω, η Ουγγρική Προεδρία ελπίζει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, τόσο ώστε τα κράτη-μέλη να συνενέσουν, να καταλήξουν σε σύμφωνη γνώμη επί τη βάση τη γνωμοδοτήσεω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, κάποια κράτη-μέλη ίσω ε, έχουν κατά νου να χρησιμοποιήσουν ε, ω βάση την αρχή πρώτα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δημόσια δεν θα έπρεπε να το λένε. Αυτό είναι προσβλητικό, είναι κόλαφο για το Κοινοβούλιο. Για το νόμο κατάργηση, για, τη, την οδηγία ε, κατά διακρι, της μεταχειρισης μεταχείρισης, Κάποια κράτη-μέλη θέλουν να ασχοληθούν, να επικεντρωθούν στο θέμα της ε, ε αναπηρίας, των ειδικών αναγκών. Θα συμφωνήσουμε κι εμείς, διότι κρίνουμε πως είναι πάρα πολύ σημαντικό η οδηγία να ε, αντιμετωπίζει το σύνολο και η προστασία από την ε, διακριτική μεταχείριση ή μάλλον ε, υπάρχουν διάφοροι λόγοι διακριτικής μεταχείρισης και εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να καταργηθεί ε, κάθε είδου διακριτική μεταχείριση λόγω φίλου, λόγω εθνικότητα κτλ. Επίσης, ε, άκουσα για αυτήν την ε, τροφό στην Ουγγαρία που τη συλλάβανε διότι έκανε τη μαμή και και εγώ το ίδιο έκανα πριν από τρία χρόνια και σοκαρίστηκα που έμαθα ότι ε, απαγορεύεται αυτό από την ε, κείμενη νομοθεσία στην ε, Ουγγαρία. Δεν πιστεύετε ότι στον τοκετό θα πρέπει να έχουν ελευθερία επιλογή οι γυναίκε. Μα είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα ω έχουν. Ευχαριστούμε κυρία Κορνέλισον. Από την Κούε τώρα η κυρία Φιγκυρέιντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα, Υπουργέ, να ε, σχολιάσω και εγώ τα ζητήματα που θέσατε. Συμφωνώ με τις ερωτήσεις ε, των συναδέλφων και δεν θα τις επαναλάβω. Θα περιοριστώ σε δύο ε, σύντομες ερωτήσεις. Πρώτον, Αυτή η πρόταση οδηγίας ε, για την άδεια μητρότητος και πατρότητος, όπως πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, για αυτό το σχέδιο, για αυτή την πρόταση οδηγίας, θα πρέπει να μας πείτε ποιες είναι ακριβώς οι προθέσεις σας και με ποιο τρόπο θα λάβετε υπόψη την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την αρχή πρόταση δηλαδή της Επιτροπής. Δεύτερη παρατήρηση. Μας ανησυχεί η κατάσταση, μας ανησυχούν οι διακρίσεις, οι διωγούμενες διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες ε, στο χώρο εργασίας ε, μας ανησυχούν οι μισθολογικές διαφορές, ε, η ανισότητα ως προς την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Επίσης, ε, οι επισφαλείς, κακώς αμοιβούμενες θέσεις απασχόλησης που συνήθως αφορούν τους γυναίκες, ο κίνδυνος φτώχειας που είναι πολύ πιο έντονος για τις γυναίκες. Η συνάδελφος Μπάουερ είδε η ήδη είπε ότι δυστυχώς ε, στην ε, στρατηγική 2020, ενώ μιλάμε για την απασχόληση, ε, δεν έχουμε συμπεριλάβει καμία αναφορά στην ισότητα των δύο φύλων. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι ανησυχητικό. Βεβαίως, πώς τίθεται το ερώτημα. Στη συγκεκριμένα, αυτά έχει πρόθεση η Ουγγρική Προεδρία να αναλάβει πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό, ε, πρωτοβουλίες που θα έχουν ε, απτά αποτελέσματα να επιχειρήσετε παραδείγματος χάρη να, να θεωρήσει το Συμβούλιο την άποψή του. Να επιχειρήσετε ε, στον προϋπολογισμό να έχουμε καλύτερα, πιο θετικά αν θέλετε αντανακλαστικά γιατί χρειάζονται και κονδύλια για να προωθήσουμε τα ζητήματα της ισότητας των δύο φύλων ε, θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης ε, των γυναικών. Σκέφτεστε κάποια συγκεκριμένα μέτρα τέλος για την καταπολέμηση των ε, μισθολογικών ε, διαφορών και για την προστασία των γυναικών από τη φτώχεια. δεν φτάνουν οι εξαγγελίες γιατί τελείω στο, φτάσαμε στο τέλος του ευρωπαϊκού έτους για την καταπολέμηση της φτώχειας και τελικά έχουμε περισσότερη φτώχεια. Το γνωρίζουμε ότι σε ένα εξάμεινο δεν μπορείτε να φέρετε τα πάνω κάτω, δεν μπορείτε να τα λέξετε όλα, το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά τρία-τέσσερα συμβολικά μέτρα θα μπορούσατε ε, να ε, εισηγηθείτε ε, τέσσερις συγκεκριμένες πρακτικές που να προωθούν τα ζητήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ε, Υπουργέ, μόλις ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Πριν ε, σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε, θα ήθελα κι εγώ να καταθέσω κάποιες απόψεις. Ε, εποφελούμε από το ότι οι διάφορες συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο θέμα της άδειας μητρότητας και της τροποποίησης της σχετικής οδηγίας. Και στο μέτρο που εγώ είμαι η στο Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα, θα ήθελα να ρωτήσω τον Υπουργό το εξή. Ποια πρόοδο μπορούμε να αναμένουμε από την Ουγγρική Προεδρία, από την παρέμβασή σας, προκύπτει ότι μειώνουμε στο ελάχιστο τις φιλοδοξίες μας. Είπατε ότι θα καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσετε τη συνοχή, να έχουμε ένα ανοιχτό και επικοδομητικό διάλογο στο Συμβούλιο κτλ. κτλ που όμως δεν θα ολοκληρωθεί ε, η Ουγγρικής Προεδρίας. Αναφερθήκατε στη δυσκολία, στην περιπλοκότητα του ζητήματος, στις ε, διαφορές που σημειώνονται από κράτο σε κράτο λόγω διαφορετικών παραδόσεων των 27 κρατών μελών, αλλά συγκεκριμένα τι μπορούμε να περιμένουμε, τι μπορούμε να περιμένουμε ότι θα συμβεί ε, κατά τη διάρκεια της δικιάς σας Προεδρίας για αυτή τη συγκεκριμένη οδηγία. Επίσης, ε, ε αν θέλετε, ε, είμαι κάπως ε, αμήχανη, ας το πω έτσι, γιατί ε, Εσχάτος ε, τροποποίησε την νομοθεσία της η Ουγγαρία και ε, σχετικά με την άδεια μητρότητας Λοιπόν, και αν το συνδέσω αυτό με τις ε, προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας, θέλετε να προωθήσετε την ε, οικογένεια, να καταπολεμήσετε ε, τη δημογραφική πρόκληση της Ένωσης, δεν υπάρχει μια ανακολουθία ανάμεσα σε αυτά που εξαγγέλλεται τώρα για την οδηγία για την άδεια μητρότητας και τους στόχους που μας εκθέτεται ταυτόχρονα, διότι Παρότι είναι αλήθεια ότι η πρόταση του Κοινοβουλίου διευρύνει επεκτείνει την άδεια μητρότητος σε σχέση με την αρχή πρόταση της οδηγίας αληθεύει ταυτόχρονα και κάτι άλλο, ότι εμείς ε, δεν είμαστε υπέρ μιας παρατεταμένης, αν θέλετε, άδεια μητρότητας, ε, υπέρ της περίοδου που, που προβλέπει η κείμενη δική σας νομοθεσία, γιατί αυτό παρεμποδίζει την επιστροφή στην αγορά εργασίας ε, και οι γυναίκες εφόσον ζητούν ισότητα θα πρέπει να έχουν και ισότιμη πρόσβαση και να επιστρέφουν ταχαίως στην αγορά εργασίας. Δεύτερον, για να τονίσουμε την ε, γενετικότητα, για να προστατεύσουμε τον οικογενειακό πυρήνα, είναι απαραίτητο και οι αδειο μητρότητας και οι άδεια πατρότητας ε, να καταβάλλονται στο ακέραιο. Ε, ε οι οικογένειες θα πληγούν οικονομικά μεσούσεις της κρίσης. Ε, ποιες προσδοκίες μπορούμε να έχουμε από την Ουγγρική Προεδρία για αυτά τα ζητήματα ε, και σε σχέση με την αρχική σας ε, παρουσίαση. Ελπίζω τώρα με τις απαντήσεις που θα μας δώσετε θα μας κάνετε ε, να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι αν θέλετε, δηλαδή να έχουμε υψηλότερες προσδοκίες σε σχέση με την, ε, ε, πρόταση οδηγίας για την άδεια μητρότητας. Έχετε το λόγο, Υπουργέ. Ευχαριστώ. Όχι. Θα, απαντήσω, λέει ο κύριος Υπουργό. Προς την κυρία Μπάουερ, καταρχάς, συμφιλίωση εργασ... επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Χαίρομαι που κατανοείτε τις προσπάθειες που γίνονται. Σας είπα, έχουμε μία ζητή προσέγγιση. Από τη μία πλευρά η αγορά εργασίας πήγαμε και στην ε, Επιτροπή του Κοινοβουλίου και παρουσιάσαμε τις ιδέες μας και από την άλλη πλευρά την προστασία των γυναικών για την οικογενειακή τη ζωή δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε ή να υπονομεύσουμε το ένα σκέλος έναντι του άλλου. Είναι γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν και επαγγελματικές υποχρεώσεις και εικονιακές και το μοίρασμα αυτών των υποχρεώσεων δεν είναι ισότιμο, δεν είναι δίκαιο. Το ξέρω ότι υπάρχουν πολλές αδικίες ε, και στο σπίτι και στην εργασία πολλές ανισότητες. Βλέπουμε γυναίκες που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν το στόχο τους να δημιουργήσουν μια οικογένεια για να μπορέσουν να προοδεύσουν στην καριέρα τους, στη δουλειά, στην επαγγελματική ζωή. Πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε προτεραιότητες και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον με συντονισμένες προσπάθειες. Υποστηρίζουμε μία αύξηση των φορέων, των οργανισμών που προσφέρουν φροντίδα για το παιδί. Ε, ό,τι και να είναι αυτοί οι οργανισμοί, οι ενώσεις, σωματεία, όλο αυτό το πλαίσιο πρέπει να ενισχυθεί της φροντίδας του παιδιού. Επίσης, ε, είμαστε υπέρ της ε, ενισχυμένης προστασίας, στήριξης των μελών της οικογένειας που είναι, είναι, φροντίζουν άλλα μέλη τα οποία έχουν ειδικέ ανάγκες ή ηλικιωμένους. Ό, όλο αυτό το πλαίσιο πρέπει να ενισχυθεί. Και αυτή η ενισχυμένη βοήθεια για της οικογένειας πρέπει να δοθεί ανεξάρτητα από το φύλλο και σε άντρες και σε γυναίκες. Θα διαβουλευτούμε με τους κοινωνικούς εταίρους. Αλλά οι κοινωνικοί εταίροι δεν θα συνυπογράψουν τη συμφωνία. Όποια συμφωνία επιτευχθεί. Προ την κυρία Τόμσον. Σας ευχαριστώ που εκτιμήσατε κι εσείς την ε, πρόθεσή μας να προωθήσουμε το θέμα της ε, βίας ε, που βασίζεται στη διάκριση των φύλων, της βίας κατά των γυναικών. Αναφέρατε επίσης ότι υπάρχουν ποσοστώσεις όσον αφορά την απασχόληση των γυναικών. Για να πω κάτι συγκεκριμένα Εξετάζοντας τις μελέτες που έχουν γίνει, μπορούμε να πούμε ότι ούτε πολίτες, ούτε κυβερνήσεις ξέρουν ακριβώς πώς, τι αποτέλεσμα έχουν αυτές οι ποσοστώσεις. Δηλαδή, δεν έχει γίνει καμία σε βάθος αξιολόγηση ε, της χρησιμοποίησης ποσοστώσεων. Ίσως αυτό είναι μια ευκαιρία να δούμε τέλος πάντων ε, αυτές οι ποσοστώσεις έχουν αποτέλεσμα και μπορούν να βοηθήσουν το ρόλο των γυναικών σε ηγετικές θέσεις, στη λήψη αποφάσεων κλπ. Ε, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε, να ενισχύσουμε τις γυναίκες όταν έχουμε καλύψει το βασικό θέμα της, ε, των ίσων ευκαιριών πρώτα να εξασφαλίσουμε ίση πρόσβαση και ίσες ευκαιρίε και μετά να δούμε αν ή όχι θα χρησιμοποιηθούν ποσοστώσει. Πιστεύω ότι πρέπει να δίνονται ίσες ευκαιρίε στις γυναίκες σε οποιαδήποτε θέση και σε οποιοδήποτε επίπεδο. Εν συνεχεία, το σχέδιο οδηγίας για την καταπολέμηση... Α, ε, τη, της κατά των γυναικών που βασίζεται στη διάκριση του φίλου. Ε, πιστεύω ότι αυτή η πρόταση θα, η δική σας πρόταση θα επηρεάσει την Κομισιόν. Όσον αφορά τώρα τη σύνθεση της ουγγρικής κυβέρνησης, δεν νομίζω ότι υπήρχε ειδική, ειδικό κάποιος ειδικός λόγος για τον οποίο όλα τα μέλη της κυβέρνησης είναι άρενες είναι μια, ένα ιστορικό συμβάν. Έτσι τέλος πάντων είναι η κατάσταση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αγνοούμε την προαγωγή των γυναικών σε κυβερνητικές θέσεις. Όπως σας είπα, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν γυναίκες σε ηγετικές θέσεις. Πιστεύω ότι είναι καθαρή σύμπτωση το ότι η κυβέρνηση της Ουγγαρίας αποτελείται μόνο από άντρες. Και όσον σε ό,τι αφορά το θέμα της, επιχει... της επικύρωσης της σύμβασης του ΟΗΕ. Και τι θα κάνουμε από αυτού. Η Ουγγαρία έχει δώσει ένα πολύ καλό παράδειγμα. Πιστεύω ότι είμαστε από, τους προ... από τις πρώτες χώρες που έχουν επικυρώσει αυτή τη σύμβαση. Αυτή τη στιγμή διαβουλευόμαστε με άλλα κράτη και αν υπάρχουν απορίες ή αβεβαιότητες ή ενδιασμοί είμαστε πρόθυμοι να, να απαντήσουμε και να διευκρινίσουμε άνθρωποι που ζουν με ειδικέ ανάγκες το θέμα αυτό είναι στην ατζέντα μας έτσι κι αλλιώ, και η επικύρωση τη σύμβαση. η άδεια, η γονική άδεια, η άδεια τοκετού και ελοχές δεν θέλουμε να πληγώσουμε τα αισθήματα κανενός και ειδικά των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Απλώς θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τη θέση μας και την προσέγγιση μας για την πρόταση της Κομισιόν. Θέλουμε να διαπραγματευτούμε στο Συμβούλιο. Αλλά σας είπα, θα αναθεωρήσουμε την αρχική πρόταση της Κομισιόν ταυτόχρονα για τη γονική άδεια. Ε, είναι λυπηρό, αλλά βλέποντας τις διάφορες θέσεις των μελών του Συμβουλίου για αυτό το θέμα, δεν νομίζω ότι ε, θα επιτευχθεί συμφωνία σύντομα. Βεβαίως θα μελετήσουμε τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Σας είπα, δεν θα το αποφύγουμε αυτό το θέμα, ούτε θα προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε. Είναι σοβαρό, θα το χειριστούμε με την πρέπουσα σοβαρότητα και μάλιστα μέσα σε μια οικονομική κρίση. Σας είπα ότι τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν το θέμα με πολύ διαφορετικές απόψεις και με μεγάλες δυσκολίες. Η επόμενη ερώτηση της κυρίας Κορνίλσεν γιατί εστιάζουμε περισσότερο στα άτομα με ειδικέ ανάγκες παρά στα σήματα των διακρίσεων του φύλου. Εγώ πιστεύω, σας είπα ότι συνεχίζουμε το έργο, το, το, τους φακέλους αυτούς της Βελγικής Προεδρίας. και ταυτόχρονα εκτός από τη διασφάλιση της συνέχειας των φακέλων αυτών τα άτομα με ειδικέ ανάγκες είναι προτεραιότητα για μας όχι μόνο για την Προεδρία αλλά και στην Ουγγαρία και γι' αυτό σας είπα ότι θα οργανώσουμε μια, ένα συνέδριο υψηλού επίπεδου που θα εστιάσει τα θέματα στην οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Η, επίσης η άλλη οδηγία 43 κάθετος 2000 που αναφέρεται στην καταπολέμηση των διακρίσεων επί τη βάση εθνότητας και αυτό θα το λάβουμε υπόψη. Για επανέρχομαι τώρα στην άδεια μητρότητος, πατρότητος τη γονική άδεια τέλο πάντων και τη διάρκεια της και την ενσωμάτωση της άδεια πατρότητος του στοιχείου της πατρότητος, της άδειας πατρότητος μέσα σε αυτές τις οδηγίες αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα διότι η οδηγία αναφέρεται στα θέματα υγείας, προστασίας, ασφάλεια των γυναικών, ε, βασικά στα θέματα υγείας κατά την, το θυλασμό, και δεν πιστεύω ότι είναι σωστό το πλαίσιο αυτό για την πρόθεση του θέματος ε, της άδεια πατρότητας. Όχι ότι έχουμε καμία αντίρρηση με το θέμα της άδεια πατρότητας, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε μια διαφορετική βάση να το ενσωματώσουμε. Ίσως αν, αν πούμε γονική, γονική άδεια, parental leave, εκεί θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στο θέμα της ε, άδεια πατρότητας. Αυτή είναι η αρχική μας προσέγγιση. Αλλά αναμένουμε βεβαίως και μία χρήσιμη συζήτηση με τα μέλη. Η κυρία Πρόεδρος επίσης με ρώτησε γιατί δεν είμαστε πιο φιλόδοξοι από ό,τι σας, σας είπα, το πρόγραμμά μας δηλαδή. Και απαντώ ότι πρέπει να επιτύχουμε μια κοινή θέση με 27 χώρες ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαμε να ήμασταν πιο φιλόδοξοι στο πρόγραμμά μας. Η Ουγγρική, το εθνικό πρόγραμμα της Ουγγαρίας και στο Εθνικό Κοινοβούλιο μας υπάρχουν προτάσεις πολύ πιο τολμηρές, πολύ πιο φιλόδοξες. Όμως πρέπει εδώ, σε αυτό το πλαίσιο, να λαμβάνουμε υπόψη και τα 26 άλλα μέλη και αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις ε, έρχονται και φεύγουν, η θέση της γερμανικής κυβέρνησης μπορεί να αλλάξει π.χ. Αλλά δεν είναι μόνο η Γερμανία που έχει πρόβλημα και άλλες χώρες, με την οδηγία δηλαδή. Εν συνεχεία, ε, θέλω να απαντήσω σε ερωτήσεις που αφορούσαν την περίπτωση αυτή της Ουγγαρέζας ΜΕΑΣ θα σας, έχω να σας πω ότι με την αφορμή της περίπτωσης αυτής συντάχθηκε ένα νομοσχέδιο το βρίσκεται τώρα προς εξέταση ε, στα χέρια των, της κυβέρνησης διότι οι τοκετοί κατοίκων δεν καλύπτονταν από καμία νομοθεσία και υπήρχαν προβλήματα σε σχέση με αυτή την επιλογή. Τώρα όμως θέλουμε να ε, εδραιώσουμε νομοθετικά αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει λοιπόν ένα νομοσχέδιο το οποίο θα περάσει από το Γκρικό Κοινοβούλιο Ελπίζουμε το νομοσχέδιο αυτό να βελτιώνει τις συνθήκες, να αυξάνει την ασφάλεια, να μειώνει τους κινδύνους και να εξασφαλίζει την αναγκαία προστασία τούτο και του κατοίκων. Σας ευχαριστούμε. Θα αρχίσουμε τώρα το δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Τώρα δεν είναι εκπρόσωπο των πολιτικών ομάδων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον Υπουργό για την παρουσίαση και για τις απαντήσεις που έδωσε. Νομίζω ότι έχουμε μια σαφέστερη ιδέα τώρα για το τι μελγενέστε στην Προεδρία σας, αλλά μας ανησυχούν ακόμη κάποια πράγματα, παρότι μίλησατε για την οικογενειακή βία, για τις μισθολογικέ ε, διαφορές και Όλα καλά και ωραία. Αυτά και όλοι χάρηκαν, όλοι οι συνάδελφοι χάρηκαν που τα αναφέρατε παρόλα αυτά. Έλειπε αυτό το θέμα της ισότητας των δύο φίλων στο αρχικό έγγραφο. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε γιατί υπήρχε αυτό το κενό. Και έτσι τίθεται και ένα ευρύτερο ερώτημα που σχετίζεται με αυτά που λέγαμε για το ότι δεν ε, υπάρχουν γυναίκες στην κυβέρνησή σας. φαίνεται να είναι πρόβλημα η συμπερίληψή τους. Είναι γενικό το ερώτημα. Κάποιες σκέψεις μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας. Δηλαδή, ε, ποιος είναι ο ρόλος των γυναικών στην κοινωνία σας, κατά τη γνώμη σας, όχι μόνο στην κοινωνία της ε, Ουγγαρίας, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη. Υπάρχουν επίσης συνταγματικές ε, προθέσεις θέσεις ε, να ε, ήδη από τη σύλληψη το έμβριο να έχει νέο, νέα υπόσταση, νομική υπόσταση ε, γιατί αυτό μπορεί να οδηγεί σε πλήρη απαγόρευση της άμβλωσης καθώς και των χαπιών για την αποτροπή της κοίησης που παίρνει κάποιος την επόμενη μέρα. ε, μήπως έτσι θέσουμε σε κίνδυνο, σε αυξημένο κίνδυνο τη ζωή των γυναικών και των παιδιών. Τι πιστεύετε εσείς γι' αυτό, το επιθυμούμε πραγματικά, το επιθυμεί αυτό η Ουγγαρία. Κάτι άλλο, επίσης ε, εγχώριο ζήτημα, ε, νομίζω ότι στο κοινοβούλιο σας ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι τάσεται υπέρ της μερικής απασχόλησης των γυναικών για να έχουν χρόνο να φροντίζουν και τις οικογένειές τους. Ε, έχουμε συζητήσει ήδη τα περί γυναικών ε, κατοίκων στο χώρο εργασίας. Ε, πιστεύετε ότι με αυτή την πολιτική θα έχετε περισσότερα παιδιά και ευτυχέστερες μεγαλύτερες οικογένειε. Θα περάσω τώρα στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Μας μιλήσατε για τη στρατηγική 2020 Ευχαριστούμε για τις απαντήσεις ε, που δώσατε, αλλά εφόσον εκπροσωπείτε την Προεδρία μπορείτε να μας πείτε τι προτίθεστε να κάνετε για να ε, διατηρηθούν οι στόχοι της διαδικασίας Βαρκελόνης ε, που σχετίζονται με τις γυναίκες. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Σνίσιν τώρα. Σας ευχαριστώ. Η σύνθεση της Ουγγρικής κυβέρνησης αποτελεί σοβαρό πράγματι πρόβλημα που σας αφαιρεί αξιοπιστία στην πολιτική αυτή για τα δύο φύλλα χρειάζεται να δει κανείς τι γίνεται και στο σπίτι του και ίσως θα έπρεπε να αλλάξει η σύνθεση της κυβέρνησης. Δεν είναι και τόσο δύσκολο το πράγμα και ελπίζω να είναι από τις προτεραιότητες της ε, Ουγγρικής ε, Κυβέρνηση, ε, η αγώνας κατά της βία ενάντια στις γυναίκες αλλά ταυτόχρονα και για τη σύνθεση της κυβέρνησης ε, συγγνώμη, την βία κατά της γυναίκας. Εδώ λοιπόν ε, θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει στην Ουγγαρία. μην έχουμε τώρα θεσμοποιημένη βία του κράτους κατά των γυναικών αυτή η βία θα είναι ας πούμε η νομοθεσία κατά τις διακοπής, εθελούσες διακοπής που είναι κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό ισχύει στη χώρα μας πούμε και τώρα στην τελευταίο ψήφισμα το Κοινοβούλιο εγγυάται στις γυναίκες ε, στο με ασφαλή τρόπο να προχωρούν σε άβλωση. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τις προτεραιότητες και μαζί με τη ε, βία κατά των γυναικών θα πρέπει να προσέξει ε, και το θέμα της βίας της έμεσης μέσω της απαγόρευσης αυτής της άμβλωσης. Ε, αυτό λοιπόν για να δούμε τα δικαιώματα των γυναικών και ο νόμος ε, κατά της άμβλωσης μειώνει τα φερή δικαιώματα από τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες και σημαίνει ότι ας πούμε το να μείνει κανείς κάποια έγκυος της αφαιρεί δικαιώματα. Αυτό σημαίνει. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα την αρχή της ισότητας. Τι θα κάνει η Προεδρία θα το εξαφανίσει αυτό να μην αντιμετωπίζονται οι διαφορετικά οι γυναίκες, οι έγκυες από εκείνες που δεν είναι ε, και σε αντίθεση και με τις γυναίκες, με τους άντρες, συγγνώμη. <clears throat> Ναι. Καλησπέρα. Θα ήθελα να χαιρετήσω την παρουσία σας εδώ και θα θέλαμε εμείς όπως και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μας που πήραν το λόγο να σας συγχαρούμε για την παρουσία σας και για το θέμα αυτό το πολύ σημαντικό. Θέματα που μας απασχολούν είναι αρκετά πέρα από θέματα εθνικής νομοθεσίας. Αλλά αυτό που αναφέρατε εσείς ιδιαίτερα με απασχολεί και νομίζω και το σύνολο της κοινωνίας. Η βία κατοίκων κατά των γυναικών, και εγώ είμαι συνσυντάκτρια μιας έκθεσης για την προστασία των θυμάτων βίας. Είναι το Ευρωόρντεν όπως λέγεται και υπάρχουν πολλές γυναίκες που θα πρέπει να βοηθούνται από τη στιγμή που γίνονται θύματα στη χώρα τους θα πρέπει και σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να τους αναγνωρίζεται αυτή η ιδιότητα του θύματος και χρειάζεται όλα αυτά να τα εξετάσουμε. Θα θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα εκ μέρους των Ευρωπαίων γυναικών και επίσης στον Υπουργό Εσωτερικών και Δικαιοσύνης σαν μέλος εγώ μιας άλλης Επιτροπής, Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών. Είχα υποβάλει ερωτήσεις αυτούς τους δύο και μου είπαν ότι θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό, με τις γυναίκε θύματα βίας, που θα παρουσιάσει το θέμα αυτό, τη δέσμη αυτή μέτρων για τις γυναίκες, θα υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά εδώ αυτό που έχει υποστηριχθεί στο Κοινοβούλιο με πλατιά πλειοψηφία χρειάζεται να περάσει σαν μέτρο και να θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι ακριβώ γνωρίζετε σε αυτό το θέμα και συνεργασία με τον Υπουργό Δικαιοσύνη και θα μπορούσε να κάνει κάτι η Προεδρία, η Ουγγρική στο Συμβούλιο ε, γιατί ξέρουμε ότι δεν υπάρχει πλειοψηφία και θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει, τι μέτρα μπορεί να λάβει ακριβώς η Προεδρία η Ουγγρική για να προστατεύσει τις γυναίκες οι οποίες είναι θύματα παρομοιας οικιακής βίας. Κύριε Δεν ακούγεστε το μικρόφωνο σας. Oh, sorry. Yes, thank you for your presentation. I must say that... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ε, παρουσίασή σας. Θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, κοινωνική πολιτική της Προεδρίας σας. Ε, έχετε πολύ φιλόδοξους στόχους να προωθήσετε τις φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές, να υλοποιήσετε την ευρωπαϊκή πολιτική για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και άλλες κοινωνικές πολιτικές. Εγώ ε, θα ήθελα να ακούσω πρακτικούς τρόπους, πρακτικά μέτρα. Και καταρχάς καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε βεβαίως ποσοστώσεις για ε, την ε, υποχρεωτική απασχόληση γυναικών. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω ποιο είναι το ποσοστό των εργαζομένων γυναικών στην Ουγγαρία ε, για τις, ε, ή, για τις γυναίκες υποψήφιες ας πούμε ε, στις εκλογές. Θα ήθελα να, ξέρω λίγο τα ποσοστά, τα εθνικά σας ποσοστά. Και ποια θα είναι η προτεραιότητα σας υπαριθμών ένα στον κατάλογο, δηλαδή Ποιο είναι το πιο καυτό θέμα με το οποίο θα ασχοληθείτε αυτό το εξάμεινο. εξάμεινο. Είναι πάρα πολύ σύντομη χρονική διάρκεια και δεν μπορείτε όλα να τα καταφέρετε. Άρα ποιο είναι πρώτο στη λίστα σας. Ευχαριστούμε κύριε Πλάμα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Υπουργό κύριο Ρέταλη. Σας άκουσα και χτες στην Επιτροπή Απασχόλησης θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Ακούστε, ε, άκουσα ακριβώς την παρουσίασή σας και διάβασα και τις προτεραιότητες ε, σας στην κοινωνική πολιτική. Και σήμερα επίσης ε, τώρα άκουσα την εισήγησή σας για τις τρεις προτεραιότητες που έχουν να κάνουν με την ισότητα των φύλων. Επιτρέψτε μου όμως σας παρακαλώ να σας υποβάλω δύο ερωτήσεις. για την αναθεώρηση του σημείου αυτού στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020 για την ισότητα των φύλων και πώς θα παγιωθεί αυτή η συμφωνία για την ισότητα των φύλων. Εσείς απαντήσατε ήδη σε μία από τις ερωτήσεις λέγοντας ότι το σύμφωνο αυτό εκεί δεν θα υπογράψουν, δεν θα συνυπογράψουν οι κοινωνικοί εταίροι και θα ήθελα να καταλάβω εγώ γιατί θα γίνει αυτό. Και ακόμα δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με τη θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Πεςτε μου κάτι. Η Προεδρία η δική σας η Ουγγρική μπορεί να μας πει ποιες θα είναι ορισμένες συγκεκριμένε πρωτοβουλίες για τη μείωση ας πούμε επίπεδου μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας και γνωρίζουμε ποιε είναι οι συνεπέπειες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κυρία Γιανακουδάκη τώρα. Ευχαριστώ. Καλά το είπατε το όνομά μου. Σωστά το προφέρατε. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Αργοπόρησα λίγο, αλλά ήμουνα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη. Εγώ ασχολούμαι τώρα με τις γυναίκες στις επιχειρήσεις και κυρίως στις μικρές επιχειρήσεις. Εχθε έγινε μια συζήτηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στην Ουγγαρία και ένα από τα θέματα ήταν τα δάνεια. Ε, Κάποιο ζήτησε από το μπατζανάκι του να είναι εγγυητή ε, για το δάνειο γιατί αλλιώ δεν το χορηγούσε η τράπεζα. Τι γίνεται με τις γυναίκες για την σύσταση επιχειρήσεων, υπάρχει διευκόλυνση δανειοληπτική. Ε, πόσο βοηθάτε τις γυναίκες επιχειρηματίες. Ε, και υπάρχει η ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών, δηλαδή συνεργασία πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στα Υπουργεία και τους μη κυβερνητικού οργανισμούς, Πρόεδρος. Μάλιστα, έτσι ολοκληρώνουμε το δεύτερο γύρο ερωτήσεων και πρωτού δώσω το λόγο στον Υπουργό. Θα ήθελα να σχολιάσω αυτό το νομικό ε, ζήτημα σχετικά με την συμπερίληψη της άδεια πατρότητας μέσα στην οδηγία. Κοιτάξτε, έχει ήδη ευρυμένη νομική βάση η οδηγία αρχικά. Ε, σχετιζόταν μόνο με την υγεία η βάση, η νομική βάση δηλαδή της οδηγίας, τώρα όμως σχετίζεται και με την ισότητα των δύο φύλων. Αυτό επιτρέπει όχι μόνο συμπερίληψη της άδεια πατρότητας αλλά και άλλα μέτρα ε, προώθησης της συμφιλίωσης ε, της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής ε, και της προώθησης της ισότητας των δύο φύλων. θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον Υπουργό. Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη να μας απαντήσετε. <clears throat> Um, Σα Σας ευχαριστώ. Θα ασχοληθώ πρώτα με την ερώτηση τη κυρίας Χάνιμπαλ. Ε, θέσατε ένα ερώτημα σχετικά με το ρόλο των γυναικών Δηλαδή, ε, αναφερθήκατε στις ίσες ευκαιρίες ε, γυναικών και αντρών. Κάτε με, είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το ζήτημα και διάφορες ερωτήσεις σχετίζονται με την κατάσταση στην Ουγγαρία και τις ουγγρικές πρακτικές. Δεν θα ήθελα να ε, μπω σε λεπτομέρειες για την κατάσταση στην Ουγγαρία, μπορώ να σας δώσω όμω κάποια στοιχεία. Μιλώντας ε, για την Ουγγαρία, ε, προσφέρουμε ε, μία επιλογή στις γυναίκες. Δηλαδή, μπορούν να επιλέξουν ένα παραδοσιακό τρόπο ζωής ή να επιλέξουν τη σταδιοδρομία τους χωρίς οικογένεια όμως. Αυτή η επιλογή οπωσδήποτε πρέπει να προσφέρεται στις γυναίκες και εμεί υποστηρίζουμε τις γυναίκες που επιλέγουν, προκρίνουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. Κρίνουμε ότι είναι η σωστότερη λύση. Ε, κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ε, στηρίξουμε ε, και τις ε, δύο πτυχές και τα δύο σκέλη χωρίς να θυσιαστεί είτε η προσωπική είτε η επαγγελματική ζωή. Αναφερθήκατε επίσης ε, στη, σε αυτό που συνέβη στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Προφανώς ε, θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Δυστυχώς, ε, λίγες μόνο γυναίκες ε, ε, απασχολούνται μερικώς, ε, παρότι υπάρχει σοβαρή ανάγκη, αν θέλετε, για γυναίκες που θα καταλάβουν τέτοιες θέσεις μερικής απασχόλησης. Έτσι θα έχουμε και μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών στην αγορά εργασίας δεν είμαστε οι καλύτεροι μαθητές, αν θέλετε, στην Ουγγαρία, αλλά υπάρχει βούληση να αλλάξουμε. Δεν ε, θέλουμε να υποχρεώσουμε τις ε, γυναίκες να επιλέγουν την μερική απασχόληση. Δεν είναι αυτή η πρόθεση της Ουγγρικής ε, κυβέρνησης. Τώρα για αυτό το συνταγματικό θέμα, κοιτάξτε τώρα εκπονείται το σχέδιο, δεν έχουμε ακόμη ε, όλες τις λεπτομέρειες και ως εκ τούτου δεν θα σχολιάσω αυτό το συνταγματικό θέμα. Ε, μου υποβάλλατε ένα ερώτημα επίσης ε, εξίσου συνταγματικού χαρακτήρα για την κυβέρνηση. Δεν θα ήθελα να το σχολιάσω. Ε, για να δω αν ε, υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση στην οποία δεν απάντησα. Η Προεδρία, η Ουγγρική Προεδρία δεν επιθυμεί να παρέμβει σε θέματα που υπάρχουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ως προς την οικογενειακή βία, Πιστεύω πως το πακέτο περί προστασίας των θυμάτων βίας είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό νομικό ζήτημα. Είπατε ότι ε, συνομιλήσατε ήδη με τον Υπουργό Εσωτερικών της Ουγγαρίας για αυτό το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα αρμοδιότητος του, όντως. Βεβαίως. Ε, οφείλουμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα για την προστασία των γυναικών, ε, διότι δεν πρόκειται για θύματα φυσικών καταστροφών. Ε, μιλάμε για την οικογενειακή βία και πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα για να βελτιωθεί η κατάσταση. Αυτά τα βήματα όμως συνεπάγονται μάλλον για να ε, καταφέρουμε να κάνουμε αυτά τα ε, σημαντικά βήματα θα πρέπει να εργαστούμε από κοινού. Πάντω συνιστά προτεραιότητα για την Προεδρία μας η καταπολέμηση της βίας που υφίστανται οι γυναίκες. Θέλουμε να αποφύγουμε τα ακραία περιστατικά. Θέλουμε ε, να αποφύγουμε τη μοιραία απόλυξη τέτοιων επεισοδίων ενδοοικογενειακής βίας, αν θέλετε itt az esélyegyenlőség κατόπιν ισότητα των ευκαιρίων, ε, ε, πρακτικές φιλικές ω προς την οικογένεια, προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρία. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα σας απαντήσω παραπέμποντάς στο πρόγραμμα της Ουγγρικής ε, Προεδρίας λοιπόν, ίσες ευκαιρίες, αναπηρίες, πρακτικές φιλικές προς την οικογένεια, όλες αυτές είναι ε, ισότιμες ε, προτεραιότητες τη Ουγγρική Προεδρία. Το βλέπετε με σαφήνεια στο πρόγραμμά μας. Αυτά είναι τα βασικότερα ζητήματα που θα συζητήσουμε στον Κοντούλο και στη Βουδαπέστη στις διασκέψεις που οργανώνουμε. θα αποδώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε όλα αυτά τα ζητήματα. Τώρα, ε, για το σύμφωνο ε, περισσότερο των δύο φίλων, δεν θέλω να ε, σχολιάσω το περιεχόμενο του συμφώνου αυτού. Πιστεύουμε είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να καλύψουμε όλες αυτές τις διαστάσεις ε, που προαναφέραμε, τις μισθολογικές διαφορές, την ε, ε, συμμετοχή στη διαδικασία λήψη αποφάσεων, ε, τι ανώτερε θέσει επιχειρήσεων, το θέμα της ε, βίας. Αυτό το σύμφωνο θα, το αναθεωρημένο σύμφωνο θα οδηγήσει σε πολιτική δήλωση των Υπουργών στο Συμβούλιο. Κυρία Γιανακουδάκη, ε, ως προς τις επιχειρήσεις, γιατί υποβάλλατε ένα σχετικό ερώτημα, Προφανώς ε, υπάρχουν κάποια μικρά βήματα που μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Η Ουγγαρία υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βέβαια δεν θέλουμε να μιλάμε για ουγγρικά, μήπως ουγγρικά ζητήματα. Για τα δάνεια μας ρωτήσατε, για τις επιδοτήσεις, για τις παροχές. Ε, δεν υπάρχουν ε, διακρίσεις, προτιμήσεις λόγω αν θέλετε. Είναι ουδέτερη η παροχή υπηρεσιών από πλευράς μας. Για τα θετικά μέτρα κατά των διακρίσεων, με ρωτήσατε, δεν ε, υφίστανται στην Ουγγαρία. Δεν ε, έχει αναλάβει τέτοια μέτρα ε, η Ουγγρική κυβέρνηση. Πολλές όμως είναι οι γυναίκες επιχειρηματίες στην Ουγγαρία. Υποστηρίζουμε τις ενώσει γυναικών, τα σωματεία γυναικών που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα. Ένα άλλο ερώτημα σχετιζόταν με τον αριθμό των ε, γυναικών που συμμετέχουν στην κυβέρνηση της Ουγγαρίας και τον αριθμό συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Δεν είναι ικανοποιητικά ε, τα ποσοστά ούτε στην κυβέρνηση ούτε στην αγορά εργασίας και θέλουμε να αυξήσουμε την αναλογία ε, Τώρα για τη συμφιλίωση ε, της ε, προσωπικής και επαγγελματική ζωής. Οφείλουμε να βρούμε σωστές λύσεις, την κατάλληλη μεθοδολογία και προφανώς ε, σε εγχώριο επίπεδο θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια μεθοδολογία για να εκριζώσουμε οποιασδήποτε ανισότητες και ανισορροπίες παρατηρούνται είτε στην Ευρώπη είτε στην Ουγγαρία. Η Πρόεδρος μας μίλησε για τη νομική βάση της ε, οδηγίας. Προφανώς θα λάβουμε αυτό που είπατε υπόψη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος, η κυρία Πλάμ έχει μία σύντομη επερώτηση, ένα σύντομο σχόλιο. Παρακαλώ, παρακαλώ και μετά θα ακούσουμε και τον Υπουργό. Um, Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ Ρέτελη, απαντώντας σε μένα μου είπατε ότι το σύμφωνο αυτό δεν θα υπογραφεί από τους κοινωνικούς εταίρους. Σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν συνυπογραφτεί από τους κοινωνικούς εταίρους θα είναι απλώς μια πολιτική δέσμευση εκ μέρους του Συμβουλίου γιατί έτσι όπως το ερμηνεύω εγώ ένα ε, σύμφωνο, ένα pact ε, σύμφωνο δηλαδή πρέπει να συνυπογραφεί από τους κοινωνικούς εταίρους ε, αλλιώς τι, τι ακριβώς θα εκπροσωπεί Ευχαριστώ Σας ευχαριστώ Δίνω το λόγο, Δίνω το λόγο να απαντήσει ο, ο Υπουργός Μα και το προηγούμενο σύμφωνο δεν είχε υπογραφεί από τους κοινωνικούς εταίρους κατά τις πληροφορίες που έχω. Καταλαβαίνω όμως ότι εσείς θέλετε να έχει κάποιο βάρος αυτό το σύμφωνο, ένα κύρος. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας και εις βάθος συζήτησης. Σας ευχαριστούμε και πάλι για όλες τις ε, πληροφορίες που μας δώσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία για την ε, Ουγγρική Προεδρία. Εμείς πιστεύουμε ότι θα, ε, είναι, θα στεφθεί με επιτυχία η Ουγγρική Προεδρία για, τον, για όλους τους Ευρωπαίους. Ευχαριστούμε. Vamos continuar com a nossa ordem de trabalhos. Θα συνεχίσουμε τώρα τις εργασίες μας. Πάμε στο επόμενο σημείο. Το 5 στην ημερήσια διάταξη για την ναι. Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για την ε, υποστήριξη της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση της Επιτροπής Γυναικών προς την καθήλια αρμόδια Επιτροπή, δηλαδή την Επιτροπή Απασχόλησης. Στις 16 η Επιτροπή Απασχόλησης θα εξετάσει την ε, έκθεση. Πρέπει και εμείς να αποφασίσουμε. Αύριο θα ψηφίσουμε. Έχουμε 29 τροπολογίες και χωρίς να χρονοτριβώ, η κυρία σενισχυνη είναι θα πάρει το λόγο τώρα για να μας ε, μιλήσει για το θέμα αυτό. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Λοιπόν, σχετικά με την ευρωπαϊκή συνεργασία στην επαγγελματική κατάργηση για να υποστηρίξω με τη στρατηγική Ευρώπη 2020, δεν έχουν ληφθεί κατάλληλα υπόψη τα θέματα της εκπαίδευσης και της μόρφωσης των γυναικών. Βέβαια, ε, καθορίστηκαν σαν μια πολύ σημαντική πρόκληση αυτά, αλλά δεν υπάρχουν ιδιαίτερε ενδείξεις για την επιτυχία της πολιτικής ισότητας στην εκπαίδευση εκπαίδευση, την κατάρτιση και πρέπει να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό, το επαγγελματικό των γυναικών, πώς θα συμπεριληφθούν στην αγορά εργασίας, όπως επίσης και την πρόσληψη γυναικών σε μη παραδοσιακά επαγγέλματα η εκπαίδευση κατάρτιση δεν λαμβάνει υπόψη τις ειδικέ ανάγκες που απορρέουν ακριβώς από τις ειδικές συνθήκες της ζωής των γυναικών και πολλές φορές οι γυναίκες πηγαίνουν προς ε, χαμηλότερα αμοιβόμενα θηλυκά επαγγέλματα και γι' αυτό υπάρχουν πολλοί άνδρες περισσότεροι που εργάζονται στην αγορά εργασία ακριβώς. Το σύστημα αυτό εκπαίδευσης και κατάστασης επαγγελματικής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ειδικέ συνθήκες για τις γυναίκες, τις φτωχές γυναίκες, τις περισσότερο ηλικιωμένε, εκείνες που έχουν γυναίκες ή προβλήματα υγείας. Εδώ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα για αυτά τα προγράμματα, δηλαδή χρειάζονται περισσότερες γυναίκες στην επαγγελματική κατάρτιση και περισσότερες γυναίκες που να εργάζονται στις μακρομεσαίες επιχειρήσεις όπως επίσης και κατοίκων και επίσης ε, επαγγελματικές συμβουλές για τις γυναίκες. Σχετικά με την στρατηγική Ευρώπη 2020 χρειάζεται να γίνει ένα ε, όλων αυτών σε συνδυασμό με την αγορά εργασίας. Εδώ εδώ κάπως ε, συνοπτικά βρίσκονται στην ε, ε, έκθεση για διοικητικού λόγους και οργανωτικούς υπήρξαν, κατατέθηκαν 29 τροπολογίες που εμπλούτησαν ιδιαίτερα αυτήν την έκθεση. Εγώ τη συμφωνώ και θα τις υποστηρίξω στην ψηφοφορία. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Κλάστα πάρει το λόγο τώρα, είναι η σχεδόν συζητήτρια του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την έκθεσή της, η οποία σε έξι παραγράφους παρουσιάζει εμπεριστατωμένα αυτό το θέμα. Και λέει όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να λεχθούν. Την ευχαριστώ λοιπόν επίσης που ανέλαβε αυτό το θέμα της ε, ισότητας, της ίσης μεταχείρισης και της ε, επαγγελματικής ανέλυξης των γυναικών στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Ε, συζητάμε χρόνια και χρόνια ίδια θέματα και επιτέλους πρέπει κάπου να καταλήξουμε. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σωστά αυτά τα οποία γράφει τα έξι σημεία. Οι 29 τροπολογίες πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν αποδεκτές σχεδόν όλες. Ε, είναι θετικέ. Εδώ όλοι προσπαθούμε να τονίσουμε την, ε, τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην επαγγελματική ζωή και στην κατάρτιση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και ε, πιστεύω ότι οι τροπολογίες εκφράζουν ειδικέ συνθήκες που επικρατούν πολλές φορές, ελλείψεις που πρέπει να διορθωθούν, ε, στερεότυπα τα οποία θα πρέπει να καταργηθούν. Υπάρχουν όλα αυτά τα στερεότυπα όπου λέει τα κορίτσια ε, καλύτερα στο σπίτι να μένουν και στα τεχνικά επαγγέλματα, στην τεχνική κατάρτιση καλύτερα να πάνε τα αγόρια, ε, ότι τα κορίτσια δεν είναι και τόσο κατάλληλα για τεχνική, ε, τεχνολογική κατάρτιση ενώ μία επαγγελματική κατάρτιση και για τα κορίτσια μπορεί να γίνει και απλά με ένα βιβλίο κατοίκων Πιστεύω λοιπόν ότι η πρόθεση της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης σίγουρα θα βοηθήσει τις γυναίκες. Ε, ας αρχίσουμε καταρχάς από την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μπορούμε να βοηθήσουμε εκεί, διότι μπορούν από εκεί να λάβουν πάρα πολλές πληροφορίες για την ε, εκπαίδευση τους, για πρόσβαση, για προγράμματα, και μπορούν μάλιστα από το σπίτι τους να, ενημερωθούν και μπορούν ε, να δουν από το σπίτι τους ε, τι μπορούν να κάνουν, τι προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν και εν συνεχεία πώς μπορούν να εξελιχθούν. Ε, όλα αυτά ενισχύουν την ανεξαρτησία των γυναικών. Οι γυναίκες δεν θέλουν ε, να εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία τους, ε, την οικονομική, λαμβάνοντας εκατομμύρια πιστώσεις, τους φτάνει ένα μικρό ποσό για να ξεκινήσουν ε, μία μικρή επιχείρηση, ίσως μία βιοτεχνία ή μία απασχόληση κατοίκων. Γενικά σας ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ την εισηγήτρια και πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε μία καλή γνωμοδότηση στα χέρια μας με καλές τροπολογίες που ανταποκρίνεται στους γενικούς μας στόχους. Έτσι πιστεύω ότι θα προχωρήσει η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρρευση των γενικών στα πλαίσια της Agenda 2020. wirtschaftlichen Spitze in der Welt. Είναι γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν να παίξουν ακόμα ένα μεγάλο ρόλο σε πολλά ε, σημεία του κόσμου. Σα ευχαριστούμε. Η κυρία Παρβάνοβα τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική της εργασία η κυρία Σένιστιν. έχει ακολουθεί ακριβώς την ίδια προσέγγιση όπως και η ομάδα μου σε αυτό το θέμα και πιστεύω ότι οι προτάσεις της προσθέτουν ε, ε, αξία στο όλο θέμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. οι απόψεις της ε, ομάδας μου και οι δικές μου συμφωνούν ε, ε, σχεδόν απόλυτα με τις απόψεις της εισηγήτριας. Πρέπει να διευκολύνουμε την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας όπως το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στην Επιτροπή μας και δι γυναικών που προέρχονται από μειονότητες, μειονοτικές ομάδες πρέπει να δώσουμε περισσότερα κίνητρα στις γυναίκες να ενταχθούν στην κατάρτιση και στην εκπαίδευση και έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία και τα προγράμματα της Ατζέντα 2020 για κίνητρα και καινοτομίες στην αγορά εργασίας έχω υποβάλει ε, προτάσεις για την απασχολησιμότητα των γεγονότων των, συγγνώμη, των γυναικών σε τομείς όπως πράσινους τομείς, μη τεχνολογικούς τομείς, σε διαφορετικούς τομείς που μπορούμε ακόμα, έχουμε ένα μεγάλο περιθώριο ενίσχυσης. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες δεν έχουν μια δίκαιη εκπροσώπηση, όχι μόνο σε υψηλές και ηγετικές θέσεις, αλλά γενικά ε, στους ε, τομείς του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ε, της υψηλής τεχνολογίας και του τραπεζικού συστήματος υπάρχει μεγάλη ανάγκη προώθησης γυναικών. Υπάρχει ανάγκη να προχωρήσουν στις καριέρες τους, να προχωρήσουν ε, να ανελιχθούν στις εργασίες τους και πιστεύω ότι με αυτή την έκθεση η Επιτροπή μας δίνει ένα ισχυρό μήνυμα ε, προς τις άλλες Επιτροπές ε, και προς το Σώμα Γενικό στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστούμε η κυρία Τσεκόβα τώρα. Ευχαριστώ. Έχω μία πάρα πολύ σύντομη παρατήρηση. Πιστεύω πως ε, δεν ενδείκνεται να έχουμε ένα κατάλογο επαγγελμάτων για τα οποία ε, ε, δεν προσφέρονται, αν θέλετε, οι γυναίκες, ότι πρέπει ε, με, σε δουλειές σε χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος να απασχολούνται οι γυναίκες. Ότι καλύτερο είναι να εμπλέκονται στην κατάρτιση και να μην ασχολούνται με τις σε εισαγωγικά παραδοσιακές δουλειές. πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα γνωμοδοτήσει η Ολομέλεια πριν προχωρήσουμε. E σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντελγκάντο τώρα εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πάρει τον λόγο. Ευχαριστώ. Πράγματι, οι παρατηρήσεις σας είναι πολύ επίκαιρες. Όταν εμείς παρουσιάσαμε αυτή την ανακοίνωση από πλευράς Κομισιόν, ήμασταν στα πλαίσια της αναθεωρήσης του πλαισίου της Κοπενχάγης, δηλαδή αναθεωρούσαμε όλο το πλαίσιο της επαγγελματική κατάρτισης και εκπαίδευσης των τελευταίων δέκα ετών. Αυτό που θέλαμε να επιτύχουμε στην αναθεώρηση είναι να καθορίσουμε μακροπρόθεσμους στόχους εν ώψη της Agenda 2020 και της στρατηγικής της, ειδικά για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ε, ίσως θεωρείτε ότι η πρότασή μας είναι υπερβολικά γενική και όχι ειδική. Ειδικά, δηλαδή δεν αναφέρεται σε θέματα της διάστασης του, των φύλων. Όμως, νομίζω ότι όταν ενισχύουμε ιδιαίτερα τον πυλώνα της συμπερίληψης όταν προτείνουμε μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν την και θα καλύψουν και τις γυναίκες, θα ενισχύσουν δηλαδή την ίση μεταχείριση μην ξεχνάτε ότι μια σωστή ισορροπία των φύλων δεν, είναι μόνο, δεν αφορά μόνο τη διάσταση του φύλου, αλλά αφορά και ειδικού στόχους για ειδικέ ομάδες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Άρα λοιπόν, ζητώντας μέτρα που θα ενισχύσουν τη συμπερίληψη και των, των ε, δύο φύλων, πιστεύω ότι προωθούμε το θέμα της διάστασης των φύλων ε, ε, λέτε ότι πέρα από τα παραδοσιακά προφίλ ε, απασχόλησης αναφύλο θα πρέπει η νέα γενιά να επιδιώξει να βρει απασχόληση και σε τομείς που δεν είναι παραδοσιακά η γυναική ή η ανδρική. Θα πρέπει λοιπόν τα παιδιά να έχουν μία ευρεία επιλογή καριέρας και δυστυχώς στην Ευρώπη, στα σχολεία, στη σχολική εκπαίδευση, ο επεγγελματικός προσανατολισμός που γίνεται για στα παιδιά δεν τους προσφέρει πολλές επιλογές. Ε, τα παιδιά υφίστανται πάρα πολλές εξετάσεις, σχολικές εξετάσεις, ε, για βαθμούς, ενώ δεν τους προσφέρεται μια σωστή εικόνα των δυνατοτήτων απασχόλησης που θα έχουν αργότερα. Πρέπει τα παιδιά να ξέρουν ποιες είναι οι επιλογές τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη διάσταση του φίλου διότι υπάρχουν, όπως είπατε, πολλά στερεότυπα, πολλές ε, αντιλήψεις παγιωμένες για τα επαγγέλματα αυτό που εκτός από τη διάσταση του φίλου πρέπει να προσέξουμε είναι οι επιλογές αυτές να είναι ελκυστικές. Πολλά επαγγέλματα δεν είναι ελκυστικά ε, για το ένα ή το άλλο φίλο και υπάρχουν πολλές παρανοήσεις για επαγγέλματα, για καριέρες όλα αυτά θα πρέπει να, να τα στοχεύσουμε στο σχολικό επίπεδο είναι στο σχολείο που το παιδί μαθαίνει για τον επαγγελματικό προσανατολισμό εγώ πιστεύω ότι η δική σας ε, συμβολή ε, προσθέτει αξία ε, στις προσπάθειές μας και ότι το έγγραφο αυτό είναι πολύ καλό για τα επόμενα δέκα χρόνια και πιστεύω ότι όλη αυτή η εργασία είναι πολύ σημαντική. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντελγάτο για τις διευκρινήσεις σας. Πολύ εύστοχα τα σχόλιά σας. Για να κλείσω το θέμα θα δώσω και πάλι το λόγο στην συγκίτριά μας για να απαντήσει, αν θέλει, ε, στις ερωτήσεις, να σχολιάσει τις παρεμβάσεις ε, ή να κάνει κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε, βάση περιπτώσει. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και πάλι για όλες τις τροπολογίες. Νομίζω ότι έτσι έχει εμπλουτιστεί ιδιαίτερα το θέμα και νομίζω ότι και αύριο θα υπερψηφιστεί όλα αυτά στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όπως ε, είπαμε ήδη αύριο θα ψηφίσουμε για αυτή την γνωμοδότηση. Θα ε, ε, ψηφιστεί στην Επιτροπή Απασχόλησης αυτή η έκθεση στις 16 του μήνα και κατόπιν το Μάιο στην Ολομέλεια θα περάσει, από την Ολο... ε, συγγνώμη, θα περάσει το Μάιο από την Ολομέλεια το σχέδιο έκθεσης. Περνάμε στο σημείο 6. Στι 9 Νοεμβρίου 2010, την προσωπία τη Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητα των ε, Φίλων στο Βελγικό Κοινοβούλιο. Είναι μια ε, καθιερωμένη επίσκεψη, αν θέλετε, γίνεται για κάθε Προεδρία. Η κυρία Σφένσον ε, μα. Ε, εκπροσωπεί εκεί και η κυρία Τόμψον θα μας ενημερώσει τώρα για τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης. Ευχαριστώ. Έγινε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και συνάντηση στο Βελγικό Κοινοβούλιο. Ε, συναντηθήκαμε με μέλη της Επιτροπής Γυναικών στο Βελγικό Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει τέτοια επιτροπή ε, σε όλα τα κοινοβουλία στη χώρα μου, Φερρυπίν, και σε άλλες χώρες. Ε, γι' αυτό και ε, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συναντούμε με μέλη της Επιτροπής Γυναικών του Βελγικού Κοινοβουλίου. Όταν συζητούμε τα θέματα ισότητας των φίλων στην Ευρώπη, πιστεύω ότι πρέπει να ε, αντλούμε την έμπνευσή μας από εθνικές ε, πρακτικές, από εθνικά βιώματα και στο Βέλγιο αυτό που με εξέπληξε είναι το θέμα του δελτίου που υπάρχει που προβλέπεται για τις οικιακές ε, βοηθούς επιχορηγούμενες, ε, δηλαδή τέτοιες ε, υπηρεσίες ε, οικιακών βοηθών. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα για την μερική απασχόληση. Εισέρχονται στην αγορά εργασίας οι γυναίκες, αλλά το ενδιαφέρον στη βελική νομοθεσία ποιο ήταν ότι ενεργοποιούνται οι γυναίκες, εισέρχονται στην αγορά εργασίας, προωθείται η σταδιοδρομία τους. Unemployed women then. Καταπολεμείται η ανεργία και οι οικιακές βοηθοί ε, πώς βρίσκει μάλλον ε, κάποια γυναίκα οικιακή βοηθό περνώντας από έναν ε, οργανισμό, από μια, ε, από μια ιδιωτική υπηρεσία εξέβρεσης οικιακών βοηθών και τι γίνεται, το βελγικό κράτος καλύπτει ένα κομμάτι της αμοιβή αν θέλετε της οικιακής βοηθού μέσω του δελτίου που σας έλεγα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το σύστημα και θα ήθελα να θεσπιστεί και σε άλλες χώρες. Θα ήθελα να ε, προσκαλέσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα μέλος της Επιτροπής Γυναικών του Βελγικού Κοινοβουλίου για να μας ε, πει όλες τις λεπτομέρειες για, αυτές τις, ε, για αυτή την πρωτοβουλία του Βελγίου. Πάντως ήταν ξεχωριστή εμπειρία. Ε, πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Τόμψεν. Κυρία Μπάουερ τώρα έχει το λόγο. Uh, Σας ευχαριστώ. Να προσθέσω κάτι κι εγώ. Ήταν μία τακτική συνεδρίαση όπως κάνουμε και σε άλλα κράτη-μέλη για να συναντήσουμε εκπροσώπους της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, το Βέλγιο δεν έχει μία κανονική κυβέρνηση, έχει μία υπηρεσιακή ε, ε, γι' αυτό λοιπόν επισκεφθήκαμε το Κοινοβούλιο και πραγματικά μας ενέπνευσε ιδιαίτερα αυτά που ακούσαμε. Αυτό το σύστημα που ανέφερε η κυρία Τόμσον είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και ε, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής για να αποφύγουμε το πρόβλημα της μαύρης εργασίας και ε, της ε, φοροδιαφυγής κλπ. Καλή ιδέα λοιπόν, πώς, μία καλή ιδέα πώς να λυθούν δύο προβλήματα με μιας, με ένα σπάρο, δύο τριγώνια δηλαδή. το σχέδιο, το νομοσχέδιο που αναφέρθηκε για την, το μοίρασμα των συνταξιδοτικών ε, δικαιωμάτων σε περίπτωση διαζυγίου μεταξύ των συζύγων. Είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον, ε, δηλαδή όταν μία γυναίκα ε, έμεινε σπίτι, δεν δούλεψε για να μεγαλώσει τα παιδιά κλπ. συνεχεία υπάρχει διαζύγιο, τα συνταξιδοτικά δικαιώματα μοιράζονται. Ε, υπάρχουν λοιπόν πολύ ενδιαφέρουσες εδώ ιδέες και θα ήταν καλό να κάνουμε μία ε, ανταλλαγή απόψεων με τους συναδέλφους από το Βελγικό Κοινοβούλιο και ίσως και από άλλα κοινοβούλια διότι εδώ στις Βρυξέλλες δεν ξέραμε, δεν είχαμε ενημερωθεί για αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες αυτά είχα να πω, να προσθέσω. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπάουερ γιατί ολοκληρώθηκε και η ημερήσια διάταξη. Ξαντλήσαμε την ημερήσια διάταξη. Αύριο το πρωί θα συνεχίσουμε. Παρακαλώ μην ξεχάσετε την ηλεκτρονική κάρτα ψηφοφορίας. Θα χρειαστεί να ψηφίσουμε με ηλεκτρονικό τρόπο με τις κάρτες. Μην τις ξεχάσετε παρακαλώ. Εσάβριον. Ε, vai começar agora <laughs> Α, τώρα ξέχασα, συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος και κλεισμένο των θυρών θα συνεδριάσουν οι συντονιστές.